Colleagues, we start. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πώς το λέμε, ναι, δεν πρέπει και να τιμωρήσουμε αυτούς που ήρθαν στην ώρα τους. Καλώς ορίσω λοιπόν όλους τους ε, παρευρισκόμενους. Παίρναμε στο σημείο 10 της σημερινής μας συνεδρίασης. Πρόκειται για μια παρουσίαση του σχεδίου δράσης Opera Vision. Είναι βασισμένο στην επιτυχημένη πλατφόρμα σχετικά με την όπερα στο πλαίσιο του προγράμματος ε, Δημιουργική Ευρώπη. Χρηματοδοτείται λοιπόν ε, το Opera Vision από αυτό το πρόγραμμα. Πρόκειται για, ένα, για μια ένωση Και θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την Audrey Junger, στην Γενική Διευθύντρια της Opera Europe και τον Λουκ το Οσόνεση. Ελπίζω να τα κατάφερα εύκολο το όνομά σας. Είναι project manager της Opera Vision. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε το project αυτό και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την ε, φτωχή παρουσία των ε, μελών. Όμως έχετε εδώ εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της Επιτροπής που έχουν έρθει για να σας ακούσουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σας δίνω λοιπόν τον λόγο αμέσως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλωσόρισμα είμαστε και ψηφιακό project και μια που έχουμε web streaming, είμαστε σίγουροι πως μας βλέπουν πολύ από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Έχουμε έρθει να σας παρουσιάσουμε το project μας σε περίπου 10 λεπτά και να σας πούμε τι κάνει η Opera Vision. Καθώς και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες ιδέες που είχαμε σχετικά με το μέλλον του προγράμματος αυτού. Φυσικά στο τέλος είναι καλοδεχούμενες ε, οποιασδήποτε ερωτήσεις. Η Opera Vision λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να φέρει την όπερα στην ψηφιακή εποχή. Πιστεύουμε στην δύναμη μιας ζωντανής παράστασης. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ευκαιρία ε, για την όπερα να μπορέσει να περάσει σε, στην ψηφιακή εποχή και να επικοινωνήσει έτσι με τον κόσμο ή τουλάχιστον με οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο ίντερνετ από το σπίτι του ή το κινητό τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.operavision.org. Μπορείτε να μπείτε κατευθείαν, δεν υπάρχουν κωδικοί, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ε, ελεύθερο περιεχόμενο. Έχουμε υπηρεσία streaming που μεταδίδει ζωντανά πολλές παραστάσεις και εσείς έχετε τη δυνατότητα να τις ε, δείτε κατόπιν ε, ζήτησης. On demand λοιπόν για παραστάσεις ε, έως και έξι μήνες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό project και όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, υπάρχει υλικό, παρασκηνιακό, προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέο σε ηλικία ακροατήριο. Και έχουμε επίσης και ένα κομμάτι του ιστοτόπου μας αφιερωμένο στους ε, νέους, στην όπερα του μέλλοντος. Και ε, η εικόνα που βλέπετε είναι από την όπερα Ξέρξης, από μια παράσταση που ανέβασε η Κόμισε Όπερ του Βερολίνου, η οποία θα μεταδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα ζωντανά. Τα project μας ε, λοιπόν έχουν έρθει στη ζωή ακριβώς χάρη στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και έχτισαν πάνω στην επιτυχία της ψηφιακή πλατφόρμας όπως είπατε και εσείς. Η Opera Europe που είναι ε, ο σύνδεσμος ε, των ε, λυρικών σκηνών ανά την Ευρώπη έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στην πρόσβαση των πολιτών σε πολιτισμικό περιεχόμενο. Υπάρχει λοιπόν πληθώρα εμπειρογνωμοσύνης, έχουμε συγκεντρώσει εταίρους από πολλούς εφορεί, από το χώρο της όπερας, του κινηματογράφου, του θεάτρου, χώρου, δηλαδή όπου αναβαίνουν παραστάσεις συνέχεια και επίσης προσπαθούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις των ε, ειδικών με τους ε, νέους δημιουργούς που, ακόμα, ε, που τώρα προσπαθούν να μπουν στο χώρο. Εδώ βλέπετε έναν κατάλογο από τους συνεργάτες μας για να καταλάβετε περί τίνο πρόκειται. Υπάρχουν ορισμένα πάρα πολύ γνωστά ονόματα στο χώρο της όπερας όπως από την Μαδρίτη, το Royal Opera House στο Λονδίνο, υπάρχουν επίσης ε, εθνικοί φορείς, το Εθνικό Θέατρο της Πράγας, το Θέατρο της ε, Φιλανδίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ε, είπε και οι συνεργάτες μου, να φέρνουμε σε επαφή νέους δημιουργούς που είναι καινούργιοι στο χώρο του streaming. να φέρουμε φορείς ε, δηλαδή οι οποίοι είναι μεν έμπειροι στο χώρο της όπερα, αλλά δεν ε, έχουν ακόμα μπει από το χώρο του streaming με την ψηφιακή εποχή. 15 μήνες μετράμε ως Opera Vision και μέσα σε αυτούς τους 15 μήνες είχαμε ανεβάσει 57 παραστάσεις Είχαμε δηλαδή στο site μας περίπου μία παράσταση να μεταδίδεται κάθε εβδομάδα. Οι, οι υπηρεσίες μας δεν προβάλλουν μόνο περιεχόμενο από τα μέλη μας, αλλά και από άλλες χώρες, από άλλες ελληνικές σκηνές όπου παρουσιάζεται ενδιαφέρον. έχουμε ανεβάσει παραστάσεις ε, που έγιναν σε χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ανεβάσαμε την, ε, και προβάλαμε την Τόσκα όταν ε, παίχτηκε στην Ρώμη. Περίπου πριν από πέντε μήνες είχαμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό. Είχαμε περίπου 200.000 200 ανθρώπους που είδαν την παράσταση από το διαδίκτυο. Επίσης προσπαθούμε να προβάλλουμε λιγότερο γνωστές παραστάσεις, λιγότερο γνωστό ρεπερτόριο. Για παράδειγμα, παραστάσεις από την Εθνική Όπερα της ε, Πολωνίας, που είναι παραστάσεις ε, λιγότερο γνωστές, εξίσου όμως ποιοτικές. Προσπαθούμε λοιπόν να προβάλλουμε έργα που δεν είναι γνωστά ε, στο ευρύτερο κοινό πέραν ε, εκείνο της χώρας τους. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες εικόνες από τα παρασκήνια της ε, παράστασης από τον πρινό της Τσεχίας. Βλέπετε εδώ τον σκηνοθέτη και τον δραματουργό που προσπαθούν να συνεργαστούν για την παράσταση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και υλικό σχετικό με την παράσταση, εκτός από την προβολή της ίδιας της παράστασης. Μέσα σε αυτούς τους 15 μήνες ύπαρξης, λοιπόν, τα κανάλια μας έχουν προβάλει παραστάσεις που έχουν δει σχεδόν 3 εκατομμύρια θεατές. Οι παραστάσεις προβάλλονται από διάφορα ψηφιακά κανάλια. Βλέπετε εδώ ότι είχαμε περίπου 2,5 εκατομμύρια θεατές ε, που είδαν έξτρα υλικό περίπου ένα εκατομμύριο θεατές που είδαν ολόκληρες παραστάσεις και γενικά προβάλλεται το έργο μας και το περιεχόμενό μας και στα κοινωνικά μέσα και σε άλλες πλατφόρμες. Η Opera Vision προσπαθεί να φέρει την τέχνη πέρα από τα σύνορα μιας χώρας. Βλέπετε εδώ πόσο, σημαντική, πόσο σημαντικό προϊόν εξαγωγής είναι η όπερα για ε, την Ευρώπη. Το κοινό αλλάζει ανάλογα με την χώρα προέλευσης, με την παράσταση που ανεβαίνει κτλ. Εδώ βλέπετε τα ποσοστά των θεατών μας αναχώρα. και η επιτυχία μας οφείλεται ακριβώς σε αυτή την συνεργασία των 29 φορέων που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της πλατφόρμας αυτής. Η συνεργασία αυτή επίσης είναι πάρα πολύ βασική για την μελλοντική μας διεύρυνση και την έβρεση νέων συνεργατών. Είναι πολύ σημαντικό για την διάδοση επίσης του πολιτισμού της όπερας αυτοί λοιπόν οι στρατηγικοί εταίροι είναι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε συχνά. Δύο από αυτούς είναι, μου είναι αρκετά προσφυλής. Είναι μια συνεργασία με το, την Ευρωπαϊκή Ένωση Οδείων, χάρη στους οποίους μπορέσαμε να προβάλλουμε τους ε, γάμους του Φίγκαρο στην πλατφόρμα μας. Επίσης, προσπαθούμε να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο e-learning μέσω της πλατφόρμας μας. Και ξεκινήσαμε λοιπόν ε, μια σειρά συζητήσεων με ε, σχολεία και ελπίζουμε μέσω της συνεργασίας αυτής να καταφέρουμε να προβάλλουμε το έργο μας και να περάσουμε στις ε, τάξεις, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να προβάλλουν το έργο μας στους μαθητές τους. Το Δεκέμβριο του 2020 το πρόγραμμα θα ε, ολοκληρωθεί και θα έχουμε φτάσει σε έναν ικανοποιητικό αριθμό θεατών. Θα έχουμε δώσει πρόσβαση σε χιλιάδες πολίτες στον κόσμο της όπερας και νομίζω ότι είναι αναγνωρισμένη η αξία του project αυτού ως προς την ε, πολιτισμική του αξία. Θεωρούμε πως η συνεργασία είναι σημαντικότερη της εμεμονωμένης προσπάθειας, γι' αυτό και στην ε, ενημερωτική μας εκστρατεία προσπαθούμε να εστιάσουμε ακριβώς σε αυτό το σκέλος της συνεργασίας και σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε κάποιες από τις ε, ιδέες μας για μετά το 2020. Είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, όμως ε, οι ιδέες που είχαμε μέχρι τώρα είναι να ε, διευρύνουμε το περιεχόμενο, να διαφοροποιηθούμε, να μην προβάλλουμε μόνο ολόκληρες παραστάσεις όπερας, αλλά και άλλες, άλλο περιεχόμενο, να διευρύνουμε δηλαδή και εμείς το ρεπερτόριό μας. Ένα από τα βασικά στοιχεία επίσης του όλου project είναι η προσβασιμότητα. Και εμείς θα θέλαμε να ενισχύσουμε την ε, διάσταση της προσβασιμότητας. Τώρα, πώς ε, μπορούμε να φτάσουμε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πώς μπορούμε να βάλουμε την όπερα στα σπίτια των πολιτών, ε, και μιλάω όχι μόνο για γεωγραφικά απομακρυσμένες, ε, απόμακρες περιοχές, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να πάνε ίδιοι στο θέατρο για να δουν μια παράσταση. Προσπαθούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τις διάφορες ε, εναλλακτικές προτάσεις. Υπάρχουν επίσης και διάφορες άλλες ε, πτυχές που δεν έχετε δει στην μέχρι τώρα παρουσίαση. Για παράδειγμα, εμείς θεωρούμε πως είναι μεγάλη ευκαιρία απασχολησιμότητας. Μπορούμε να, δώσουμε, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης στο χώρο της όπερας. τα διάφορα θέατρα μπορούν να αποκομίσουν γνώσεις το ένα από το άλλο και να τις μεταδώσουν στο, σε ένα νεότερο κοινό. Καθώς και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά. Τώρα με την, ε, στην ψηφιακή εποχή έχουν την δυνατότητα να χαράξουν τη δική τους ψηφιακή στρατηγική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και με χαρά θα σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν εντυπωσιακή επισκόπηση. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι εγώ δεν γνωρίζω πολλά για την όπερα, αλλά ε, θεωρώ πως ε, αποτελεί πραγματικά στο το Opera Vision μια εξαιρετική ευκαιρία. Και, την, ε, και πέρυσι είχαμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητας γενικότερα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εδώ έχουμε και ένα παράδειγμα ως προς το τομέα στον οποίο μπορεί η ψηφιοποίηση να συμβάλλει στην προσβασιμότητα του πολιτισμού και ειδικότερα στις ε, αγροτικές ε, περιοχές. Δηλαδή, θα λέει κανεί ότι θα ήθελα πολύ να μεταβώ στη Ρώμη για παράδειγμα να παρακολουθήσω μια όπερα, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση από αλλού, έστω και από το να παρακολουθήσει μια τέτοια όπερα. Άρα λοιπόν θεωρώ πω αποτελεί πραγματικά αυτό το παράδειγμα ένα πραγματικό υπόδειγμα ως προς το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιοποίηση ε, και για, την, ε, ε, για αυτόν τον τομέα των τεχνών. Και όπως είπατε και εσείς, μπορεί να αποτελέσει μια λύση για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή άτομα τα οποία διαβιούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και κατά συνέπεια δεν μπορούν να μεταβούν εύκολα σε ένα σημείο που υπάρχει παραστασία Οπότε σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για αυτό το project και στη συνέχεια και ε, απευθύνομαι τώρα στους συναδέλφους, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήματα ή σχόλια. έλεγα τρίπλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Εγώ είμαι ε, μου αρέσει πολύ η όπερα. Εντάξει, μπορεί να μην έχω πολύ εμπειρία, αλλά πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ ορισμένε όπερες Και εκείνο που θα ήθελα ε, να μάθω, ε, για το οποίο θα ήθελα να με ενημερώσετε περισσότερο, είναι προσπάθειες που κάνετε να έρχεται πιο κοντά στους νέους γιατί βέβαια δεν είναι ε, τόσο εύκολο όσο για παράδειγμα η μουσική pop ή άλλα ε, μουσικής αλλά γνωρίζετε και την ε, σχετική ε, ταινία η οποία αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα δηλαδή καλών συνθετών οι οποίοι έγιναν γνωστοί παγκοσμίω και εκεί δόθηκε η ιδέα το πώς είναι δυνατόν να ε, έρθουν σε επαφή ακριβώς με αυτούς τους ε, συνέντες προκειμένου ακριβώς να γίνουν πιο ενεργοί σε αυτό το με σε περισσότερες πρόσβασεις για τους νέους. Οπότε ε, θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι κάνετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες ούτω ώστε να επιτύχετε αυτήν την μεγαλύτερη πρόσβαση στους νέους. Και μετά αυτό το ζήτημα της καλύτερης προσαρμογής της όπερα στην ε, ε, ψηφιακή ε, μετάβαση και τη σχετική αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης. ποια είναι τα μοντέλα τα οποία έχετε κατά νου όταν κάνετε τη σχετική αναφορά. Παρακαλώ. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μια εμπειρία για τα παιδιά το να συμμετέχουν σε μια δημιουργική διαδικασία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το project την ένα ε, περιορισμένο αριθμό σχολείων γιατί ακριβώς δεν έχουμε βέβαια και άπειρο προσωπικό. Ε, δημιουργούμε όμω μοντέλα με τα οποία θα μπορούν οι καθηγητέ να ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα ε, στα σχολεία χωρί να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Γιατί βέβαια τα σχολεία δεν έχουν ε, το απαραίτητο προσωπικό για να στέλνουν τα άτομα στις διάφορες όπερε μαζί με του μαθητέ. Οπότε είναι κάτι το δύσκολο. Άλλωστε υπάρχουν και μεγαλύτερες έκταση χώρες όπου για παράδειγμα εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη πόλη για παράδειγμα οι όπερες. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένε όπερε οι οποίε εστιάζουν στο Μάντσεστερ ή στο Λίτζι σε κάποια συγκεκριμένη πόλη, χωρί να αποστέλνουν δηλαδή του θεάτρου του σε, ε, σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν με αυτά τα μοντέλα προσπαθούμε να μεταβιβάσουμε, να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία ω εργαλείο στα χέρια των διδασκάλων μέσα στι αίθουσε διδασκαλία. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, κάνουμε μία σειρά από πράγματα. Αυτό που θεωρούμε εμεί είναι ότι οι διάφορες όπερες έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιες αυτή την διαδικασία. Ε, πριν από κάποια χρόνια ήταν ε, ε, πολύ εξαρτημένες οι όπερες από την γραφειοκρατία και Και βλέπαμε ότι ε, συχνά έξω από ε, πολλές όπερε ε, υπήρχαν μπαν τηλεοπτικής αναμετάδοσης τα οποία έχουν υποκατασταθεί σιγά σιγά με αυτό το νέο μοντέλο και βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε μία, έναν τρόπο εργασία τώρα, ο οποίος είναι λιγότερο επαχθής για τον οποίο χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι χωρί βέβαια να μειώνει την ποιότητα. Δηλαδή πάντοτε χρησιμοποιείται ο ίδιο εξοπλισμό, απλώ χρειάζονται λιγότερα άτομα. Άρα λοιπόν ενθαρρύνονται οι όπερε να ε, συνεργάζονται με έμπειρου ε, ε, παραγωγού στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία και να μην χρειάζεται να βασίζονται σε κανάλια ραδιοτηλεοπτικά. οι εταίροι μας τώρα προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις που κάνει η με διαφορετικούς τρόπους. Ε, για παράδειγμα, κάποιοι αξιοποίησαν αυτά τα κονδύλια για να προβούν σε γενικές συμφωνίες με τις ε, όπερες τους, πράγμα το οποίο έναν έξυπνο τρόπο επένδυσε αυτών των κονδυλίων ειδικότερα τη σήμερα ημέρα καθώς ε, γνωρίζουν όλοι ότι ε, ποια είναι η σημασία των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης και κατά συνέπεια θεωρούν ότι εμείς αποτελούμε έναν τρόπο ακριβώς για να μην έχουν περισσότερα έξοδα στην προσπάθεια που κάνουν για να γίνουν πιο ψηφιακές. Για να ε, είμαι ειλικρινής, αντιμετωπίζουμε κάποια περισσότερα προβλήματα με τους εκδοτικούς οίκους, γιατί Προφανώ στο πλαίσιο των δικαιωμάτων των ε, δημιουργών ε, οι δημιουργοί θα πρέπει να λαμβάνουν τα, τα, κατάλληλα έσοδα. Αλλά βέβαια είναι συζητήσιμο το τι ακριβώς είναι δίκαιο. Ε, και έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο με σε διάφορους εκδοτικού οίκους αφού η εικόνα στα διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφοροποιείται. Όμως ε, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα εδώ γιατί υπάρχουν ε, κάποιες ε, από τις αξιώσεις που κάνουν οι οποίοι είναι πραγματικά υπερβολικές και θα πρέπει να μετριαστούν λίγο. Σας ευχαριστώ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα όσα είπατε. Γνωρίζω ότι για την εξέλιξή σας από το προηγούμενο πρόγραμμα έχω δει επίσης ε, τέσσερα θέατρα όπερας από την Ιταλία που συμμετέχουν και δεν υπάρχει μόνο το European School αλλά και το Europa Canto συμμετέχει και πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 50.000 παιδιά στην Ιταλία έρχονται σε επαφή μέσω ε, μια ειδική οργάνωση που έρχεται σε επαφή με το σχολείο να κατανοήσουν την όπερα και να κάνουν και τις δικές τους παραστάσεις στα θέατρα. Είπατε ήδη κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε πώς θα επενδύσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι ένα θέμα αλφαβητισμού για την ε, όπερα, αλφαβητισμού των παιδιών, αλλά και να γνωρίσουν και καλύτερα τι υπάρχει στα παρασκήνια. Δηλαδή, πώς εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Εσείς σκοπεύετε περισσότερο να αναμεταδίδετε ε, την τις παραστάσεις της ε, όπερας, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τα θέματα πνευματικής διοκτησίας και τα λοιπά, ή σας ενδιαφέρει να γνωστοποιηθεί περισσότερο πώς γίνεται μια σκηνοθεσία πώς ακριβώς απασχολούνται οι άνθρωποι με την όπερα. Δηλαδή έχει ε, και διδακτική χρειά ε, η πρωτοβουλία σας ε, ή απλώς σας ενδιαφέρει μια προσέγγιση των παιδιών με την όπερα. Δηλαδή τι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ η απάντηση να είναι σύντομη γιατί αλλιώς δεν θα μας τάσει ο χρόνος. Νομίζω είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι είναι πιο σημαντικό, γιατί και τα δύο τα προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ένα project όπως το Opera Vision είναι μεγάλη ευκαιρία εκμάθησης για τις όπερες και έχουν εκπαιδεύσει προσωπικό για αυτέ τι νέε θέσει εργασία που δεν υπήρχαν πριν. Αλλά ταυτόχρονα, αν ναι, ναι, δεν υπάρχει και κοινό να το παρακολουθήσει, δεν έχει νόημα. Εργαζόμαστε λοιπόν και στα δύο επίπεδα. Και η Opera Europe οργανισμός οργανισμό επικεντρώνεται στο επαγγελματικό σκέλο, ενώ έχουμε μια ειδική ομάδα για την απεύθυνση στο κοινό. <laughs> <laughs> Σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Σούνεκ έχει ε, τώρα το λόγο, τον οποίο θα ήθελα και να καλωσορίσω θερμά εδώ στην Επιτροπή ε, γιατί αντικαστά τον ε, κύριο Μπόγκταν Βέντα, τον συνάδελφό μας, ο οποίος ανέλαβε βέβαια τα χρέη δημάρχου και έτσι μας εγκατέλειψε. Έχετε το λόγο συνάδελφε για δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς διαδέχομαι τον κύριο Βεντάκη. Ήδη ήμουν βουλευτής, αλλά ήμουν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος για 10 χρόνια. Βέβαια, ασχολούμαι και με τα θέματα πολιτισμού. Θα μιλήσω τώρα πολωνικά. No Mm, Έχω παρακολουθήσει αυτό το project με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να ενθαρρύνω την πρόεδρο της Επιτροπής να δει πώς ε, εργάζονται τα προεδρία στα διάφορα κράτη-μέλη που εκπροσωπούν τα κοινοβούλια και την Κομισιόν, ε, τα γραφεία δηλαδή ε, γιατί δεν δημοσιοποιούν ε, αυτά τα προγράμματα. Θα μπορούσαν να, ε, να αναφέρουν στους πολίτες θέματα που τους ενδιαφέρουν. Και έχω και μια ερώτηση. Υπάρχει ένα σύστημα εγγραφής ή μπορούν οι θεατές να αφήσουν τα σχολιά τους, μπορούν να πούν τι πιστεύουν για την παράσταση. Εγώ προέρχομαι από την ε, Κρακοβία, στην Νότια Πολωνία και η όπερα της Κρακοβίας έχει συνάψει μια συμφωνία με την ε, όπερα της Νέας Υόρκης και μια μεγάλη αλυσίδα κινηματογράφων. Δηλαδή υπάρχει μια εκστρατεία για να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να πάνε στον κινηματογράφο και να παρακολουθήσουν ζωντανά τι παραστάσει τη όπερα από τη Νέα Υόρκη. Αυτό μπορεί να είναι ένα άλλο τρόπο ε, για να αυξηθούν οι συμπράξει. Και τώρα θα κάνω ένα σχόλιο στα σου είπατε εσείς. Πολλοί άνθρωποι συνδέουν την όπερα με την Πολωνία. Αυτή είναι κάπως δυτική απάντηση. Δηλαδή, ουσιαστικά, πολλές φορές παραμελούν την Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να απαντήσω αμέσω σε αυτό, γιατί μάλλον δεν ήμουν σαφή. Αυτό που εννοούσα είναι ότι η συγκεκριμένη παράσταση, που είναι υπέροχη, ήταν ιδιαίτερη. Και αυτό ακριβώ ε, μας ε, ευχαριστεί, ότι έχουμε ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι γνωστό ε, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό και εμείς το φέρνουμε πιο κοντά Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι ακριβώς να προβάλλουμε ε, λιγότερο γνωστά έργα σε ευρύτερο κοινό. Και συμφωνώ απόλυτα ότι τον τελευταίο καιρό ό,τι μέσο προβάλλεται πρέπει να είναι και διαδραστικό. Πρέπει να φτάνει στο ακροατήριο και να λαμβάνουμε ε, τις ε, εντυπώσεις του και στην όπερα μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό. Αυτό όμως προσπαθούμε να αλλάξουμε. Κάθε φορά που, μεταδίδεται, που αναμεταδίδεται μάλλον μία παράσταση, βλέπουμε πως υπάρχει μία κοινότητα που παρακολουθεί το web streaming, που σχολιάζει και όπως ε, σας είπαμε και πριν, είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στα κοινωνικά μέσα. Και συμφωνώ απόλυτα πως χρειάζεται να διασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, ε, σχολείων. Έτσι μαθαίνουμε και έτσι μαθαίνει ο ένας θεατής από τον άλλο και έτσι διαδίδεται ε, η γνώση και ο πολιτισμός. Φυσικά και αυτό δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπίλντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν, δόθηκαν απαντήσεις, δεν θα τα ξαναπώ. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστη αυτή η πρωτοβουλία. Ξέρουμε ότι στι αίθουσε των θέατρων και των οπερών είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε τους νέους ε, παρόλες τις ε, ελκυστικές τιμές. Ε, όμως, ίσως κάποιοι πεπισμένοι να επισκεφτούν αυτές τις ιστοσελίδες. Μπορούμε βέβαια να περιμένουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα προκαλέσει και επιθυμία στους νέους. Μην διστάσετε μάλιστα να στοχεύσετε και σε ακόμη πιο νεαρό κοινό. Από ό,τι βλέπω δεν ε, θα είναι, δεν θα θέτει και πολλές απαιτήσει. Ε, ε, δεν ε, έχει αναφερθεί τίποτα για τις περιοχές της Βρετάνης, όμως ε, και εμείς θέλουμε να μην προσφέρουμε ένα τυποποιημένο πολιτισμό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε στους συμπολίτε μας ε, το αίσθημα ότι ανήκουν στο ίδιο πολιτισμό. Από την άλλη το να καθιστούν ε, προσβάσιμο αυτό το πολιτισμό σημαίνει ε, ότι θα προωθούμε την Βέβαια λυπάμαι που είναι μόνο σε τρεις γλώσσες η ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα του Facebook είναι μόνο στα αγγλικά. Θα ήταν ε, κρίμα το Opera Vision ε, να έχει περισσότερους επισκέπτες ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο παρά από την Πολωνία και ίσως θα ήταν καλό να το διορθώσετε αυτό για να έχετε μεγαλύτερη απεύθυνση στο κοινό και να είναι πιο ελκυστική η ιστοσελίδα σας. Σα herzlichen ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε. Ε, Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε εκ του σύνεγγυ τι δραστηριότητέ μα. Έχετε δίκιο. Είναι σε τρει γλώσσε. Ε, το αρχικό project είναι σε έξι γλώσσε. Και βέβαια έχουμε δει ότι ακόμη και οι επισκέπτες από την Πολωνία επισκέπτονται το αγγλικό site και ε, τελικά ίσως ε, δεν αξίζει να δώσουμε χρήματα για να μεταφράσουμε το περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες. Ε, πολωνικά, Ιταλικά, Ισπανικά έχουμε και τουλάχιστον το 85% των επισκέψεων ε, είναι στις τρεις ε, κύριες γλώσσες. Βέβαια, αν είχαμε πρόσθετο προπολογισμό και περαιτέρω χρόνο θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε ανάπτυξη περαιτέρω της ιστοσελίδας και ίσως για τις, ε, θα μπορούσαμε να καλύψουμε για κάποιες ασιατικές γλώσσες ή τα αραβικά. Ja, vielen, σας ευχαριστούμε θερμά που ε, ήσασταν σήμερα εδώ και μας ε, παρουσιάσατε αυτό το εξωτερικό, εξαιρετικό συνομή, project γιατί και για μας είναι πολύ ενδιαφέρον ορισμένες φορές να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα κονδύλια που επενδύουμε εδώ στον δημιουργικό τομέα και πραγματικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, θαυμάσια project τα οποία ελοποιούνται με αυτά τα κονδύλια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα εδώ και μας παρουσιάσατε αυτό το project. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, ε, το οποίο σχετίζεται άμεσα και με τα όσα συζητήσαμε μόλις ε, τώρα, δηλαδή την ε, εξέταση των τροπολογιών σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027. Η συγκέντρια είναι η συνάδελφος Σίλβια Κώστα. Έχουμε 586 τροπολογίε οι οποίε έχουν υποβληθεί και στι 20 Φεβρουαρίου θα γίνει μια ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μα σε σχέση με όλε αυτέ. Ενώ η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα ψηφίσει στι 2 Μαρτίου. Τουλάχιστον αυτή είναι προ το παρόν ημερομηνία. Δίνω όμω τώρα το λόγο στη συνάδελφο Κώστα για να μα ενημερώσει ω προ το πού βρίσκονται τα πράγματα. Νομίζω ότι αντί για τους σκιώδεις μάλλον έχουμε τη σκιά των συγητών εδώ. Δύο συναδέλφους, βλέπω. Τέλο πάντων, τρεις συναδέλφους έχουμε συνολικά. Είναι μικρός ο αριθμός, λυπάμαι για τη μικρή παρουσία. Η Ευρω... Δημιουργική Ευρώπη αποτελεί ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της Επιτροπής μας, μαζί με το Εράσιμους και άλλα. Είναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα και στους πολίτες ε, και γι' αυτό εμείς ε, ζητήσαμε διπλασιασμό του προϋπολογισμού στο να φτάσουμε στο 2,8. Αυτή τη συζήτηση βέβαια θα την κάνουμε στο τέλος. Και όπως είπες Πέτρα, ο γενικός στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου και της εγγενούς αξίας του πολιτισμού, της δημιουργικότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας ε, των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Με το πρόγραμμα αυτό, και αυτό το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί κάναμε και κάποια βήματα προς το μπρος που τα ζητήσαμε στην εφαρμοστική μας έκθεση. Δίνεται δηλαδή μεγαλύτερη, διάσταση, μεγαλύτερη προσοχή στην ε, διεθνή διάσταση, στη συνεργασία με διεθνή προγράμματα και στην αξιοποίηση των ε, διάφορων ε, τρόπων εφαρμογής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, είχαμε περίπου 568 τροπολογίες συμπεριλαμβάνονται εδώ και οι 104 από τη δική μου έκθεση. Ήδη συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο με τους σκιώδεις εισηγητές. Εκεί εγκρίναμε 28 συμβαστικές τροπολογίες και εργαζόμαστε και σε τεχνικό επίπεδο και έχουμε προχωρήσει γιατί ήδη 60 τροπολογίες ε, είναι υπό τεχνική έγκριση και θα έχουμε και άλλε δύο συνεδριάσεις, 30 Ιανουαρίου, 12 Φεβρουαρίου και θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε την προθεσμία του Φεβρουαρίου για την ψηφορία στην Επιτροπή. Θέλαμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να καταρθώσουμε σε πρώτη ανάγνωση να ολοκληρώσουμε το κείμενο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ευχαριστώ και την Γραμματεία για τη βοήθεια. Τώρα το πρώτο σημείο εμείς Πέρα από ότι συμφωνούμε με το γεγονό ότι πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό, αυτό συνδέεται και με το περιεχόμενο. Γιατί σίγουρα έχουμε ενωπιόν μα ένα πρόγραμμα και με αυτό συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες που αυξάνει τι δράσεις της Δημιουργικής Ευρώπης, κυρίω σε ό,τι αφορά το σκέλος του πολιτισμού. Αν δεν έχουμε λοιπόν επαρκή προπολογισμό, αυτό είναι απογοητευτικό ε, για τους επαγγελματίε του κλάδου και επίσης ε, έχουμε και το σημαντικό θέμα της συνεργασίας. Σήμερα φτάνουμε στο 12-13% ε, του ποσοστού επιτυχίας. Έτσι λοιπόν εδώ θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, ε, θα έλεγα ότι θίγουν όλα τα θέματα. Θα αναφερθώ σημείο προς σημείο. Ε, κάναμε ήδη, όπως σας είπα, μια εργασία για τους πρώτους 28 συμβιβασμού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρξει η αναγνώριση ενός νέου στόχου μεταξύ των νέων στόχων των γενικών στόχων. Έχουμε δύο γενικού στόχου του κειμένου τη Κομισιόν Προσθέσαμε και εμείς ε, το στόχο του αγγενούς αξίας του πολιτισμού και το να υπάρχει ελευθερία έκφρασης ε, του πολιτισμού και το πόσο συνεισφέρει για την ε, προσωπική και κοινωνική εξέλιξη. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Δεύτερο, για τους ειδικού στόχους. Συμφωνήσαμε ότι τρεις ειδικοί στόχοι που προβλέπονται ανασκέλος. Έχουμε προσθέσει το θέμα της κινητικότητας και έχουμε λάβει και πολλές τροπολογίες και το θέμα της συλλογής των δεδομένων και της ανάλυσης δικτών ως οριζόντιοι στόχοι μεταξύ των τομέων. Επίσης, σημαντικό είναι να προσθέσουμε την ευρωπαϊκή προσταμένη αξία. Δεν υπάρχει αυτό περιέργως. Αλλά και σε ό,τι αφορά και τα περιεχόμενα, δηλαδή να υποστηρίξουμε και τα αφηγήματα που έχουν ευρωπαϊκή κουλτούρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος του πολιτισμού, έχουμε 49 τροπολογίες. Ήδη έχουμε σχεδιάσει 8 συμβαστικές τροπολογίες και αφορά μια νέα προτεραιότητα, δηλαδή την προώθηση της έκφρασης της καλλιτεχνικής έκφρασης ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων. Υπήρξε μεγάλη συμφωνία για το θέμα αυτό, για το νέο πρόγραμμα για την κινητικότητα, την συμμετοχή των πολιτών, ο αντίκτυπος ε, για την ε, κοινωνική διάσταση της συμμετοχής, ε, επίσης μεγαλύτερη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και κατόπιν έχουμε λάβει βάση κάποιων τροπολογιών, κυρίως από το Άλτενα, ένα συγκεκριμένο σημείο για την ε, εφαρμογή της ικανότητας και την εμπλοκή των επαγγελματιών αλλά και των καλλιτεχνών και την, ε, διεθνή, την ενίσχυση της διεθνούς διάστασης ε, των σχεδίων αλλά και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Εγώ έχω ενισχύσει και κάποιες τροπολογίες που θέλω να βελτιώσουν τις προτάσεις Κομισιόν, δηλαδή ενισχύοντας τη γραμμή για τη μουσική, για την ε, κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών και την δυνατότητα να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέσω και της σφραγίδας αριστείας. Το κάναμε αυτό και σε άλλους κανονισμούς για το σκέλος media. Έχουμε 20 ευτεροπολογίες, έχουμε διάφορους συμβεσμούς εδώ σε ό,τι αφορά ε, και την πολιτιστική κληρονομιά που είναι κάτι καινούριο. Θα πρέπει να προστατεύεται και η πολιτιστική κληρονομιά και τα αρχεία, τα οπτικοακουστικά αρχεία και τα ψηφιακά αρχεία και θέλουμε να προωθήσουμε τον οπτικοακουστικό κλάδο. Μου φαίνεται σημαντικό εγώ έλαβα, αλλά ήδη το είχαμε βάλει στο παράρτημα, αλλά το τονίσαμε στο κείμενο τώρα, ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής. Δεν υπήρχε αυτός ο όρος πριν. Ξέρω ότι η Κομισιόν εκπονεί ένα νέο ορισμό για ε, τις ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, όμως υπάρχει αυτή η αρχή μέσα στο κείμενο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο για τα media είναι η σύνδεση με τις νέες προβλέψεις ε, της οδηγίας για τα οπτικοκουστικά μέσα που προβλέπει επενδύσεις ε, στην εθνική παραγωγή κτλ. Κατόπιν ε, συμφωνήσαμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνσέφεραν στη συνέχεια για το να αναφερόμαστε συγκεκριμένα στα είδη που πρέπει να προωθηθούν, παραδείγματο χάρη, βιντεοπαιχνίδια, ε, κινούμενα σχέδια και άλλα. Έχουμε εδώ 24 συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και δίνουμε και μεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο ε, του European Help Desk και σε όλες τις ε, δραστηριότητες και στις καινοτόμε προσεγγίσεις που πρέπει να υποστηρικτούν διατομεακά. Ε, ένα θέμα επί το οποίο θα πρέπει να βρούμε καλύτερο ορισμό είναι το θέμα των κριτηρίων αξιολόγησης. Θέλουμε να έχουμε πιο πιατικά κριτήρια για να εξετάσουμε τα προγράμματα. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ένας πιο συγκεκριμένος συνδυασμός στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών για την αξιολόγηση, που σήμερα είναι ανεπαρκή. Και έχουμε υποβάλει και κάποιες προτάσεις στο κείμενο. Βέβαια, ακόμη δεν έχουμε βρει συμφωνία. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολλές τροπολογίες πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση για τη δημιουργία του μηχανισμού εγγύησης. Εδώ έχουμε το Invest EU και έχουμε αναφέρει τους στόχους, στην ιδιαιτερότητα του τομέα και νομίζω ότι κάναμε βήματα προς τα μπρος, γιατί στην πρώτη πρόταση Κομισιόν είχαμε απλώς ένα τίτλο, αλλά δεν είχαμε λεπτομέρειες για τις ε, λεπτομερείς ε, δράσεις το παραρτημά 99 τροπολογίες ε, στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών θα βρούμε και τις κατάλληλες συμβαστικές τροπολογίες υπάρχει ε, ένα θέμα που πρέπει ακόμα να συζητήσουμε και με την Κομισιόν και ευχαριστώ για την προσοχή που έχετε δώσει εμείς καθώς δεν έχει δοθεί απαραίτητη προσοχή στο παρελθόν στο τμήμα του πολιτισμού Γι' αυτό διατηρούμε την ομολογία 58-32 ε, που υπήρχε στο κείμενο της Κομισιόν. Η πλειοψηφία των ομάδων συμφωνεί για αυτήν την υποδιέρεση του προπολογισμού στο εσωτερικό. Αν και υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση, εμείς ε, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την αλλογία, προς τα εκεί Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο που πρότεινε και υπάρχουν διάφορε τοπολογίε που πηγαίνουν προ αυτήν την κατεύθυνση αλλά με ε, διαφορετικού τρόπου. Δηλαδή να υπάρχει μία ε, ποσοτική και ποιοτική συλλογή δεδομένων για του τομεί πολιτισμού και τη δημιουργία. Εγώ έχω μιλήσει για ένα παρατηρητήριο. Κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν κάτι διαφορετικό για το θέμα αυτό. Συμφωνούμε μεν αλλά προτείνονται διαφορετικέ λύσει, και γι' αυτό πρέπει ακόμα να βρούμε μια ισορροπία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Λοιπόν, θα τελειώσω τώρα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Κάτι άλλο σημαντικό είναι το εξή. Πολλοί συνάδελφοι συμφώνησαν και θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο παράρτημα για να προσδιορίσουμε καλύτερα τις δράσεις, γιατί εκεί είχαμε μόνο τίτλους στο κείμενο της Κομισιόν. Μιλώ για συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένε δράσει και προτεραιότητε που πρέπει να αναφέρονται στο παράρτημα για του διάφορου τομεί. Η απόλυτη καινοτομία ε, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πέντε νέους τομείς όπου παρεμβαίνουμε λεπτομερέστερα. Προτείνουμε κατεξουσιοδότηση πράξης ε, σαν ε, εργαλείο διακυβέρνησης, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο να καθορίζει προτεραιότητες και στόχους θα γίνει σεβαστός κατά τη διάρκεια της επταετίας, αφήνοντας βέβαια και την απαραίτητη ευελιξία στα τίσια προγράμματα εργασίας. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Λυπάμαι που απουσιάζουν κάποιοι συνάδελφοι, αλλά εκπροσωπούνται κάποιε ομάδε και του ευχαριστώ πολύ. Γιατί βλέπω ότι τουλάχιστον ε, έχουμε εδώ τρει-τέσσερι εκπροσώπου των ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάρουν το λόγο και οι συζητητέ, ξεκινώντας με τον κύριο Σούνεκ. Για τρία λεπτά το πολύ, παρακαλώ.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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουνικ και η Μαρτίνα Μίχελς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την Σίλβια Κώστα. Θεωρώ πως ήδη έχουμε φτάσει αρκετά μακριά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε εξάλλου. Γι' αυτό δεν θέλω να επαναλάβω κάτι που ήδη έχει υποθεί στην Επιτροπή. Για μένα είναι επίσης ε, σημαντικό το ότι καταφέραμε να αναγνωρίσουμε την αξία του πολιτισμικού προϊόντος ε, και την θέση του στον ε, πολιτισμικό διάλογο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που αυτό φαίνεται στο κείμενο. Ταυτόχρονα είναι εξίσου σημαντική η ενίσχυση της δημιουργικής βιομηχανίας η προώθηση του πολιτισμού με την ε, μορφή υποδομών. Έχουμε καταθέσει μια σχετική τροπολογία, μάλλον πρόκειται να καταθέσουμε μια σχετική τροπολογία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα σας ζητήσω να την στηρίξετε. Τώρα νομίζω πως ε, με την συνεργασία και το καλό πνεύμα συνεργασία θα οδηγηθούμε σε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το λέγω έχει Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες, είναι αλήθεια αυτό. Δεν θα επαναλάβω βέβαια αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Η εγγενής αξία του πολιτισμού είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντική και σε πολιτικό επίπεδο, όπως είπε η Μαρτίνα Μίχελ αλλά και ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Σούνιξ αυτά που είπε. Να σταθώ όμω λίγο περισσότερο στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προπολογισμό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για οτιδήποτε κάνουμε. Είναι επίση σημαντικό και ο καταμερισμός ε, το, της χρηματοδότησης. Χρειάζεται να γνωρίζουμε ε, τα διαθέσιμα κονδύλια, διότι μόνο έτσι θα ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με, τις, ε, με τα διάφορα σκέλη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Και αναφέρθηκε ήδη πως υπάρχει το νέο πρόγραμμα «Η μουσική Κίνη την Ευρώπη». Είναι μια διαφορετική προσέγγιση, απευθύνεται στους νέους. Γι' αυτό δεν θέλουμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλες ε, ήδη από την αρχή όλε τι δυνατότητε του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν έχουμε περιθώριο να αλλάξουμε την κατανομή των κονδυλίων και τα προβλήματα που έχουμε θα τα λύσουμε μόνο με πρόσθετη χρηματοδότηση. Και το ξέρω πως ακούγεται βαρετό όταν επαναλαμβάνομαι ξανά και ξανά, όμως αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Αν θέλεις καλύτερο, πιο ποιοτικό δημοσιογραφικό σκέλος, ε, πιο ποιοτικό ρεπορτάζ, τότε χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Αν θέλεις να φτάσεις σε περισσότερο κοινό, ιδιαίτερα όταν έχεις μικρά προ... μικρής κλίμακας προγράμματα όπως το Opera Vision, χρειάζεσαι χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα του προπολογισμού και της κατανομής του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα καθορίσει τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση προτού μάθουμε τι ακριβώς χρηματοδότηση θα έχουμε. Αυτό το είπα και στον Επιτροπό Ναύρατσι, στο Στρασβούργο, την περασμένη εβδομάδα. Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε κονδύλια από το ΕΦΣΥ ή τα διαρθρωτικά ταμεία και για την ευελιξία και για υποδομές διότι και τα δύο είναι σημαντικά για τον πολιτισμό. Πρέπει όμως να επιμείνουμε στην ουσία, δηλαδή τον προπολογισμό για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Να σταματήσω όμως εδώ, διότι είπα εξάλλου ότι είναι σημαντικό για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Αυτό που αναφέρω δηλαδή επανειλημμένα εδώ στο Κοινοβούλιο και ειδικότερα στην Επιτροπή μας ασκούνται μεγάλες επίεσεις ε, και δείχνει να έχει δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός ε, εδώ ε, στο Κοινοβούλιο σε σχέση με το ποιος καταλήγει πρώτος σε μια συμφωνία στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Όμω θεωρώ πω αυτό δεν ωφελεί τη θέση μα. Ουσιαστικά δηλαδή υπονομεύουμε τη διαπραγματευτική μα θέση ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί προτού συμφωνηθούν τα πάντα. Οπότε αν αρχίσουμε εδώ τώρα και ακολουθούμε κάποιε περίεργε ε, πρακτικέ, υπομονωπεύοντα ή ε, καταστατικώντα σε κάθε περίπτωση ε, τους, τον κανονισμό μα εδώ, θεωρώ πω είναι σφαλμένο. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε εμεί ω Επιτροπή, να ολοκληρώσουμε κανονικά την πρώτη μα ανάγνωση με του αριθμού που εμεί αποφασίζουμε εδώ στην Επιτροπή μα και από εκεί και μετά με την έναρξη τη νέα ε, θητείας του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα έχουμε λάβει πλέον τα οριστικά νούμερα να καταλήξουμε σε κάτι, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα προτού εμ, έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα οικονομικά στοιχεία. Αλλά πραγματικά το να κάνουμε εδώ τώρα κάποιες ε, ε, κρυφές ε, προδιαπραγματεύσεις ή προσυμφωνίες νομίζω πως ουσιαστικά υπονομεύει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω πως αυτή τη στάση λοιπόν του να είμαστε ξεκάθαροι θα πρέπει να την ακολουθήσουμε τόσο σε σχέση με το Erasmus όσο και σε σχέση με το Creative Europe και το ανέφερα στον πρέσβη την προηγούμενη εβδομάδα γιατί είχε ξεκινήσει να μου αναφέρει κάτι τέτοιο. Μπορούμε λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε με κάποιε προκαταρκτικέ διαπραγματεύσει και να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων σε σχέση με κάποια βασικά σημεία. Όχι. Για μα δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια ε, διαδικασία γιατί ή φοβούμαστε ότι θα υπάρξουν περικοπέ των κοντιλίων. Και αν είναι να υπάρξουν περικοπέ ε, κοντιλίων, τότε σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κανένα είδου εκ των προτέρων συμφωνία ε, ή οτιδήποτε παρόμοιο με το Συμβούλιο και νομίζω πως αυτή είναι η θέση στην οποία θα πρέπει να επιμένουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Κυρία Μπίλτε, έχει το λόγο. Ε, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ έχω τοποθετηθεί μέσω των τροπολογιών μου για το φάκελο αυτό. Επομένως, θέλω να πω ότι εκτίμησα πολύ τον αρμονικό τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε όλοι. Εγώ θέλω να πω όμως ότι αισθάνθηκα να έχω αποκλειστεί κάπως από αυτόν τον αρμονικό τρόπο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Απευθύνομαι στην Επιτροπή. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Αρνητικό νεύμα από την Επιτροπή. Οπότε, ο λόγος σε ένα Σίλβια. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για την διαθεσιμότητά σας να βρούμε ένα κοινό σημείο ισορροπίας. Να απαντήσω σε κάποια επικριτικά σημεία, κύριε Σόνικ. Όταν αναφέρεστε στον όρο παρατηρητήριο, βλέπετε, βάζουμε χρησιμοποιώντας και τους υφιστάμενους φορείς. Δηλαδή υπάρχει το GRC, το Κοινοερευνητικό Κέντρο, ή υπάρχουν και άλλες δυνατότητες χωρίς να δημιουργήσουμε ένα νέο κτίριο. Απλώς ε, θέλουμε έναν υπεύθυνο φορέα γιατί αυτό λείπει εντελώς. Και αυτό συμβάλλει στην αδυναμία του τομέα. Γιατί μας ε, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας ε, το παρατηρητήριο του Στρασβούργου. Δεύτερον, θα βρούμε συμφωνία και για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε μόνο ποσοτικά στοιχεία και να μιλάμε για τον αριθμό των θεατών και τον αριθμό των περιστάσεων. Δεν μπορούμε όμω ε, να βλέπουμε μόνο αυτά τα στοιχεία. Για την ε, συνάδελφο, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί. Χέλγα, έχει θέσει δύο σημαντικά θέματα. Τα έφερα και στην αρχή και τα έφερε και η πρόεδρο. Αναμφισβήτητα, η θέση μα είναι να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε ένα κείμενο του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Δεν υπάρχει ε, καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όμως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες άλλες εναλλακτικέ ε, για διάφορα άλλα project, ε, το χάρη για την ηθαγένεια. Βλέπουμε ότι ζητήθηκε από τη Λίμπε να πάμε στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που τελικά δεν βοηθάνε για να κατανοήσουν και οι άλλοι απ' έξω τη θέση μας. Αυτό είναι μια παρένθεση βέβαια. Χέλγα, έχεις δίκιο και το είπα εγώ και τις προάλλες. Αναμφισβήτητα η φιλοδοξία αυτού του προγράμματος που καλύπτει πολλές νέες δράσεις, κυρίως στο σκέλος του πολιτισμού, σχετίζεται πάρα πολύ από τον προπολογισμό. Γιατί αυτό εμείς είπαμε ότι με το δικό μας προπολογισμό και τώρα ε, βέβαια υπερασπίζομαι όλο το κείμενο σίγουρα θα ενδιαφέρει, αλλά αν βρεθούμε απέναντι στο σημερινό νούμερο, σίγουρα όλες οι νέες δράσεις και για τη δημοσιογραφία ή για τη μουσική, ο σχεδιασμός, η πολιτιστική κληρονομιά, κινδυνεύουν να είναι υποχρηματοδοτούμενες οι δράσεις αυτές. Τώρα εγώ βασίζομαι εδώ στη δική μας πρόταση προπολογισμού και ελπίζω να υλοποιηθεί. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι το θέμα της εσωτερικής κατανομής των πόρων. Γιατί αν δούμε ότι δεν αρκούν οι πόροι ή θα τροποποιηθεί η εσωτερική κατανομή μεταξύ των τομέων ή θα πρέπει να φτάσουμε στο δικό μας νούμερο. Ξέρουμε ότι είναι ανοιχτό αυτό το πρόβλημα. Πάντως εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε και να προσφέρουμε στο επόμενο κοινοβούλιο ένα κείμενο από το οποίο δεν θα μπορούν να απομακρυνθούν και να σεβόμαστε και τόσα είπαμε στο Γκέτεμπουργκ, δηλαδή ε, η Ευρώπη ε, να έχει ένα τομέα πολιτισμού και δημιουργίας. Και αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δεν θα προχωρήσει ούτε καν το ευρωπαϊκό project. Και συμφωνώ και για το θέμα του ανταγωνισμού της οπτικοκουστικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ και κλείνουμε εδώ τη συζήτηση αυτή σε ό,τι με αφορά. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ θερμά Σίλβια και εσένα και τους και όλους και σας εύχομαι καλή επιτυχία και κάτι συνέχιση των εργασιών σας. Ε, βέβαια ότι θα τα καταφέρετε και βέβαια η ψηφοφορία μας θα λάβει χώρα εδώ στις 20 Φεβρουαρίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη σημερινή μας συνεδρίαση. Στη συνέχεια θα λάβει χώρα και η συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών συγγνώμη, των συντονιστών, διορθώνει αμυνέτρια και η επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα θα λάβει χώρα στι 4 Φεβρουαρίου ανάμεσα στι 3 και στι 6.30 το απόγευμα. Σα ευχαριστώ όλου για την παρουσία σας σήμερα εδώ και καλό βράδυ σε όλου. Καλό απόγευμα. Σα ε, παρακαλώ οι συντονιστέ να παραμείνουν μέσα στην αίθουσα εφόσον παρευρίσκονται ήδη εδώ. Και οι να έχουν έναν εκπρόσωπο εδώ. Το ταχύτερο δυνατό ευχαριστεί η Πρόεδρος και τους ε, διερμηνείς για την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ.